πρόεδρο της Επιτροπής και είπα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφαλείας με θέμα θρησκευτικέ ελευθερίες ε, και πολιτιστική διαφορετικότητα. Πρώτος ομιλητής ο κύριος Κούρκουλας εκ μέρους ε, της κυρίας Άστον. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη. Τα ζητήματα που αναφέρονται στο σχέδιο ψηφίσματος ε, του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικά και ε, άπτονται πολλών ζητημάτων. Εκ μέρου τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Βαρονισάστων, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη σημερινή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεχίσει την προώθηση και υπεράσπιση σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο τη αξία στι οποίε βασίζεται. Την το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Τον Ιούνιο του 2012 υιοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο άνδρες και γυναίκες ζητούν να ζουν με ελευθερία, αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε ανοιχτέ και δημοκρατικέ κοινωνίε. Ε, που διέπονται από ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Συνεχίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες ε, για την υπεράσπιση της οικουμενικότητας αυτών των αξιών. Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της στρατηγικής μας του 2012 ήταν η υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις θρησκευτικέ ελευθερίες και πεπιθήσεις που αξιοποιούνται πλέον στις εξωτερικές μας πολιτικές. Αυτές οι κατευθυντήριε γραμμές έχουν αξιοποιηθεί στις αντιπροσωπείε μας ε, και διαπραγματεύσεις με τρίτε χώρε, διμερό και πολυμερό για την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφή ε, ε, διακρίσεων βάσει πεπιθήσεων ή θρησκευματο. και επιπλέον σε κοινή δήλωση της 20 Σεπτεμβρίου 2012, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και εκπρόσωποι τριών οργανώσεων Ισλαμικής Συνεργασίας, Αφρικανικής Ένωσης και Αραβικής Λίγκας, η Αραβικής Ένωσης, ε, ζήτησαν Αραβικού Συνδέσμου, ζήτησαν ε, συνεργασία ακριβώς για την ε, προβολή της σημασίας της ε, των θρησκευτικών ελευθεριών και καταδίκασαν οποιαδήποτε μορφή θρησκευτικού μίσου. Οι θρησκευτικέ πεπιθήσει έχουν αξιοποιηθεί για την τροφοδότηση ε, του μίσου ε, και τη αντιπαράθεση. Και μάλιστα αυτό σε όλο τον κόσμο ζήτησαν από, από όλους τους πολιτικούς ηγέτες, είτε αυτοί είναι θρησκευτικοί είτε κοσμικοί, να προασπίσουν ακριβώ αυτές τις ιδέες. Εμείς θέλουμε, την, είμαστε υπέρ πάντα της ε, ανοχής ε, και ε, του διαλόγου. Είπατε εκπρόσωπος Κάθριν Άστον και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ειδικό τη εκπρόσωπο, τον κύριο Λαμπρινίδη, έχουν προωθήσει αυτό το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα και έχουν καταδικάσει την, ε, τις διακρίσεις ε, βάσει υπεπιθύσεων ή θρησκεύματο όπου συμβαίνει αυτό είπα ότι εκπρόσωπος ε, έχει εκφράσει πολύ ρητά την ε, καταδίκη της ε, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία όπου στις 27 Μαρτίου καταδίκασε τις στοχευμένες δολοφονίες πολιτών βάσει εθνικότητας και θρησκείας και εξέφερε την ανησυχία της για την ευαλωτότητα κάποιων μειονοτήτων που γίνονται θύματα αντιπίνων. Ενώ τονίζουμε τη σημασία της, ε, ε, της καταπολέμησης ε, κάποιων αρνητικών φαινομένων, στηρίζουμε και τις προσπάθειες που γίνονται από κάποιες αρχές για την προώθηση του διαλόγου και κάποιων πρωτοβουλειών. Εμείς έχουμε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες διαπολιτισμικού και διαθεσκευτικού διαλόγου σε ένα πνεύμα ανοιχτό, συνεννόησης και αμοιβέ κατανόησης και στο πλαίσιο της UNESCO, του, της Συμμαχίας των Πολιτισμών του ΟΗΕ, ε, του Ιδρύματο Ανελίν και της διαδικασία τη Κωνσταντινούπολη. Με την υπογραφή ε, του Μνημονίου Κατανόησης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης UNESCO του 2012 ξεκίνησε μια ενισχυμένη συνεργασία. Μοιραζόμαστε κοινού στόχου για την ενδυνάμωση τη δημοκρατία, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υπεράσπιση τη ειρήνη και την ενίσχυση τη αηφόρου ανάπτυξη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ισχυρότερη πολυμερή συνεργασία. Η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα τη UNESCO συμπεριλαμβάνουν στήριξη για την κατάρτιση νέων ε, ε, προσφύγων από τη Συρία στην Ιορδανία. Το μέσο διευκόλυνση για την ε, στήριξη πρωτοβουλειών που αφορούν τον πολιτισμό σε 13 χώρε. Αντίστοιχε πρωτοβουλίε στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο και τη διατήρηση και αποκατάσταση ε, στην χειρογράφων στον Τιμπουκτού ή άλλων ε, ε, μνημείων στην Συρία. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό τμήμα της όλης συζήτηση γιατί είναι και πολύ σημαντικό τμήμα της πολιτικής μας της αναπτυξιακής. Πάντα υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συμπερίληψη, την ποικιλομορφία την πολιτισμική, για την ε, ενδυνάμωση της ειρήνης και την αηφόρα ανάπτυξη. Ο ρόλος ε, της UNESCO στην ε, αντίστοιχη αυτή πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντικός. Θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι φορέας ανάπτυξης και η στήριξη προς τον πολιτισμό είναι στήριξη προς την ανάπτυξη στις 5 Μαΐου θα γίνει στη Νέα Υόρκη μία εκδήλωση που διοργανώνεται από την UNESCO ακριβώς για τον ε, σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ ανάπτυξης και πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται και την ποικιλομορφία των πολιτισμικών εκφράσεων. Εμείς διδραματίσαμε πολύ σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση το 2005 ε, της ε, σύμβαση τη UNESCO και ένα από του κύριου στόχου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στι σχέσει μα με τρίτε χώρε είναι η στήριξη της ε, ανάπτυξης της πολιτικής ε, πολιτισμού και ε, η προώθηση ακριβώς αυτής της σύμβασης. Υπό την ηγεσία της Επιτρόπου Βασιλείου και με την ενεργό συμμετοχή της αντιπροσωπής μας στο Πεκίνο, η Κίνα έγινε η πρώτη πιλωτική περίπτωση που σχεδιαγραφεί ακριβώς τον ρόλο του πολιτισμού στην διπλωματία μεταξύ λαών και στην αμοιβαία κατανόηση στο πλαίσιο των εξωτερικών μας σχέσεων. Ο Γενικό Γραμματέα τη ε, ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ο κ. Πιαβλημό, πρόσφατα όρισε στο γραφείο του συντονιστή πολιτισμικών θεμάτων και υποθέσεων, που ε, εργάζεται συμπληρωματικά με τα κράτη-μέλη για την προώθηση τη συνεργασία και σε αυτό το τομέα. Ο συντονιστή τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση συνάπτει επαφές με μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών ε, στο διεθνές ε, πολιτισμικό σκηνικό. Η πρωτοβουλία της περισσότερη Ευρώπης, την οποία στηρίζει και η κοινωνία των πολιτών, επίσης δρά ακριβώς ε, στην διαβούλευση μεταξύ αρκετών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Σύνδεση με τα Πολιτισμικά Ινστιτούτα ήταν επίση στην πρώτη γραμμή αυτή τη συζήτηση. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου δικαίω τόνισε τη σημασία τη καταπολέμηση, τη πάλη μάλλον κατά τη θανατική ποινή. Έχουμε μία πολύ ισχυρή θέση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ε, καμία τέτοια διαφορά δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει, ε, διαφορά απόψε δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμα στη ζωή. Έχουμε καταδικάσει δημοσίω και συνεχίζουμε να το κάνουμε την χρήση της θανατικής ποινής υπό οποιασδήποτε συνθήκες και σε οποιαδήποτε χώρα. Συνεχώς τονίζουμε και στους διαλόγους μας με τρίτες χώρες είτε μέσω της ε, δημόσιας διπλωματίας, ακριβώς ε, τη βαναυσότητα αυτής της ε, απαρχαιωμένης μορφής, της απαρχαιωμένης ποινής. και αναλαμβάνουμε δράση οπουδήποτε και οποτεδήποτε εφαρμόζεται αυτή η πεπαλαιωμένη ποινή. Και μάλιστα υπάρχει και ψήφισμα για πάυση των εκτελέσεων που έχει υπογραφεί και θα συνεχίσουμε ε, στην ε, Γενική Ολομέλεια του ΟΗΕ αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Κούρκουλα, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ σήμερα την υπάτη εκπρόσωπο και περιέλαβε πράγματι στην ομιλία του όλα όσα ζητούνται ε, ήδη με την έκθεση αυτή. είναι γεγονός ότι πολλές φορές οι πολιτιστικές διαφορές και οι θρησκευτικές διαφορές έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία για την ανακίνηση του μίσους για την ανάπτυξη της θεωρίας ότι ποτέ δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα σε αυτά τα θέματα και κυρίως για μισαλόδοξες προσεγγίσεις. είναι γεγονός ότι στις μέρες μας υπάρχουν θρησκευτικές μειονότητες παραδείγματος χάρη που υποφέρουν σε διάφορες χώρες και χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι και εβραίοι και μπαχάοι δηλαδή ένα πλήθος ε, ανθρώπων που έχουν μια διαφορετική άποψη ακόμα και μέσα στην ίδια θρησκεία. Επίσης χρησιμοποιούνται ομάδες επιθετικές στα ζητήματα της θρησκευτικής διαφορετικότητας και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ευρώπη η οποία έχει τις αρχές και αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη σύμβασης ε, του συμβουλίου της ευρώπης των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη πλευρά με πολλές από αυτές τις χώρες πρέπει να συνεργαστεί. πρέπει να συνεργαστεί στο εμπόριο πρέπει να συνεργαστεί στα θέματα ανάπτυξης. το ερώτημα είναι πώς χρησιμοποιεί η ένωση αυτά τα εργαλεία για να μπορέσει να μεταφέρει όχι τη δική της πολιτιστική άποψη ή πολιτική άποψη αλλά κυρίως για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου θα συγκεραστούν όλες οι απόψεις και θα μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινά σημεία. Και βεβαίως αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να απολαύσουμε περισσότερες δημοκρατικές ελευθερίες σε πολλές χώρες και πολλά καθεστώτα. Ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πράγματι ε, λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο ενώ ταυτόχρονα η κοινοβουλευτική διπλωματία παίζει τεράστιο ρόλο καθώς και οι πολιτιστικές σχέσεις εφόσον μάλιστα όλα αυτά βασίζονται στην εκπαίδευση γιατί η εκπαίδευση είναι το σωστότερο εργαλείο. μέσα σε αυτό το πλαίσιο ειδικό ρόλο έχει το θέμα της ισότητας των δύο φύλων το πώς μεταχειρίζονται δηλαδή τις γυναίκες πάρα πολλά καθεστώτα μέσα στο πλαίσιο ανάδειξης των δίθεν πολιτιστικών διαφορών που καταλήγουν σε μυσαλλοδοξία γιατί τελικά καμία θρησκεία στα βασικά της γραπτά δεν περιλαμβάνει τη μυσαλλοδοξία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για όλη την εργασία που έγινε στα διάφορα θέματα όλο αυτό το διάστημα γιατί είναι η τελευταία μου ομιλία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σήμερα το οποίο εγκαταλείπω και θέλω να ευχαριστήσω και το προεδρείο του κοινοβουλίου καθώς και όλους τους συναδέλφους και να ευχηθώ τα πράγματα να προχωρήσουν πιο γρήγορα να γίνουν περισσότερα και σημαντικότερα για τη δημοκρατία την ελευθερία την ανάπτυξη και την άνοδο της νέας γενιάς για ένα κόσμο διαφορετικό και καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί κυρία Γκάμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να χαιρετήσω αυτά που είπε η κυρία Γιαννάκου. Όχι μόνο για την τελευταία της παρέμβαση στην Ολομέλεια όπως είπε, αλλά κυρίως για το ανοιχτό της πνεύμα, για την αποδοχή πολλών θέσεων της δικής μου ομάδος στην έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Θέλουμε αυτές οι αρχές να είναι οικουμενικές και πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εξυπηρετούν αυτές τις πολιτικές και να πριτανεύουν φυσικά και στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες που συνάπτουμε σε πολυμερές επίπεδο, σε επίπεδο εμπορίου κτλ σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτημένο όπως σήμερα η αμοιβαία γνώση, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών έχει ιδιαίτερη σημασία. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτές οι παγκόσμιες και οι οικουμενικές αρχές να οδηγήσουν σε μια συνένεση όλων γύρω από αυτές τις αρχές που είναι ακριβώς και η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή ξενοφοβίας, εξτρεμισμού, μυσαλλοδοξίας και μίσους Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά παραμένουν σημαντικέ και συνεχεί προκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε έναν κόσμο ο οποίο δεν είδε να τελειώνει η ιστορία όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν εθνοτικές, οικονομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν θα πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης για να οξύνουν την ανθρώπινη εκμετάλλευση, την ένδια, όπως βλέπουμε στην κεντροαφρικανική δημοκρατία όπου οι διαφορετικές ε, θρησκείες και οι χρήστους ουσιαστικά συγκαλύπτουν πολύ βαθύτερα εσωτερικά προβλήματα. Στον αγώνα λοιπόν αυτό είναι απαραίτητο να μην ξεχάσουμε ότι ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία που βασίζεται στο θρησκευτικό φανατισμό είναι μια και που είναι μια από τις πιο διαστρεβλωμένες μορφές εξτρεμισμού είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει και μέσα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι ο Ισλαμικός ε, εξτρεμισμός έχει περισσότερα θύματα μουσουλμάνους από άλλες θρησκευτικέ ε, ε, κοινότητες. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να ακούμε τους σκοταδιστές οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία σαν όπλο. Είναι απαραίτητο ως κοινοβουλευτική εμείς να τονίζουμε την ανάγκη προστασίας των μειονοτήτων στην Μέση ε, Ανατολή που την χάνουν θύματα εξτατιών στοχευμένων εναντίον τους ενώ είναι μειονότητες οι οποίες έχουν ζήσει εκεί επί χιλιάδες χρόνια και <clears throat> ενισχύουν τις χώρες που βρίσκονται. Αλλά έχουμε και τις κοινότητες των μουσουλμάνων που είναι το κύριο θύμα του εξτρεμισμού και της βίας στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο λόγος και κλείνω κύριε Πρόεδρε Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αγωνιστεί για την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου, για τους μηχανισμούς αποτελεσματικής πολυμέρειας και να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία των προσπαθειών στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να σταματήσει η ατιμορρησία. Ευχαριστούμε κύριε Γκόμες. Ακολουθεί ο κύριο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εδώ και δεκαετίες δεν έχουν γίνει τόσες καταδιώξεις χριστιανών όπως τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει στο Πακιστάν, στο Ιράκ και στη Συρία. Στις χώρες αυτές και ιδίως στη Συρία και το Ιράκ. Είναι ολόκληρες κοινότητες χριστιανών που είναι από τις παλιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο, αυτές έχουν ουσιαστικά εξολεθρευτεί ή αναγκαστεί να μεταναστεύσουν. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία εμεί είμαστε συνυπεύθυνοι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να προστατεύσει αυτούς τους, χριστιανισμού, τους χριστιανούς, όχι μονάχα τους άθεους και τους αγνωστικιστές, αλλά και τους χριστιανούς αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει ανυπεράσπιστοι. Υπάρχει το σημείο 30, το οποίο μιλάει για την αρχή της αμοιβαία ερεσιμότητας. Αλλά χρειάζεται να σκεφτούμε πώς αυτό το πράγμα εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Τουρκία. Πού υπάρχει αμεβαιότητα. Η Τουρκία υποστηρίζει ομάδες δολοφόνων που έχουν στραφεί εναντίον χριστιανών, έχουν δράσει σε, στα σύνορα της Συρίας και έχουν ουσιαστικά εξαλείψει χωριά Αρμενίων στην Τουρκία. Η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει κάπου αλλού. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία έχει κάνει την πρώτη μεγάλη γενοκτονία το 1915 κατά των Αρμενίων, μια μεγάλη καταδίωξη κατά των χριστιανών. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία γίνονται είναι ουσιαστικά από την Τουρκία, είναι ένα φιλοσυκής για τους Ουαχαμπίτες και αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε με τίποτα. Κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ήρθα σε επαφή με διάφορες θρησκευτικέ κοινότητες και πάντα υπερασπίστηκα την ελευθερία διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ε, ειδικά ε, σε ψηφίσματα κατεπήγοντα που, συζητάμε κάθε πέμπτη απόγευμα. Έχω πάντα καταδικάσει τη βία εναντίον θρησκευτικών κοινοτήτων. Είτε είναι Εβραίοι, Βουδιστές, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, τα μέλη των κοινοτήτων αυτών δεν έχουν θεμελιώδη δικαιώματα μόνο και μόνο γιατί είναι μέλη μιας κάποιας θρησκευτική κοινότητας με μοναδικό κριτήριο αυτό. Ε, διάφοροι κρατικές αρχές αποπειράθηκαν να κλείσουν ε, εκκλησίες ή τις κατέστρεψαν ή υπήρξαν διώξεις ε, χριστιανών στο Πακιστάν, Φερρυπίν, ε, λόγω των νόμων ε, περί βλασφημίας. Πέρα από τις σχετικές αντιδράσεις, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνεκτική στρατηγική, μια συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε την, τις άπειρες μορφές της Γι' αυτό πιστεύω ότι η κυρία Γιαννάκου μίλησε πάρα πολύ σωστά και θα πρέπει ε, η εξωτερική μας πολιτική να διαπνέεται από αυτές τις αρχές. Ε, αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Ξέρω ότι συχνά τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διαφωνούν ε, για τέτοια θέματα. Αλλά θα πρέπει γύρω από κάποιες βασικές ιδέες και αρχές όλοι να συμφωνήσουμε και να προωθήσουμε κάποιες σαφείς δράσεις. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Γιαννάκου ότι οι πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές πολύ συχνά χρησιμοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο ως πρόσχημα για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πηγές ε, πόλωσης και συγκρούσεων και βίας εξτρεμιστικής. Αρκεί να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αιγυρία. Τη Δευτέρα στο Αμπουτζάν ε, έγινε μια επίθεση με πάρα πολλά θύματα. Πάνω από 150 άτομα χάσαν την ζωή τους ε, από τις αρχές του 2014 ε, λόγω της βίας του Μπόγκο Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε φυσικά και η στρατηγική μας θα πρέπει να είναι συνεπής, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι θα πρέπει συστηματικά να τονίζουμε ότι η μυσαλόδοξη ερμηνεία οποιασδήποτε θρησκείας που επιτρέπει τη βία και την καταστολή δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες και την καθολικότητα των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η κυρία Λούτσεβα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Υποστήριξα το ψήφισμα για την ε, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της πολιτιστικής και σκεφτικής ποικιλομορφίας. Εμείς εκπροσωπούμε διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά εκπροσωπούμε και τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να έχουμε κοινέ και σαφείς αρχές για να χτίσουμε τις ε, σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί χώρες με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική ταυτότητα, με διαφορετικές αξίες, έχουμε το σοβαρό καθήκον να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική η οποία να μην παραβιάζει την ε, κυριαρχία των κρατών μελών και να προστατεύει παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πολιτιστική ποικιλομορφία, τις διαφορές, τις σκεφτικέ διαφορές. Συχνά αυτές οι διαφορές έγιναν πηγή εντάσεων και συγκρούσεων και αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Αντί να μιλάμε για ε, ανοχή, μιλάμε για εξτρεμισμό, ξενοφοβία, που είναι φαινόμενα τα οποία δεν είναι καινοφανή στην Ευρώπη. Τα έχουμε συναντήσει και τους περασμένους αιώνες στην Ευρώπη και θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία μας σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τέτοιους κινδύνους. Η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε μια σταθερή δημοκρατία, διεθνή συνεργασία και επιθυμία για επικοδομητικές λύσεις για όλα τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την, τις αξίες οι οποίες αντιβαίνουν στη δημοκρατία. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική καθορίζει και προδικάζει την εξέλιξη βασικών περιοχών του πλανήτη. Αν εμείς ε, δράσουμε σωστά θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία για μελλοντικέ γενιές σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Υποστήριξα πολλές από τις ε, ιδέες της, ε, του ψηφίσματος. Έχουμε, ας πούμε, Σύριους ε, πρόσφυγες. Ε, υπάρχει το πρόβλημα της ξενοφοβίας που δεν το έχουμε ξεπεράσει. Στη χώρα μου, όταν αυξάνονται οι πρόσφυγες, έχουμε ποικιλόμορφες αντιδράσεις. Ε, χάρη, Βλέπετε και τις διαφορές στην Ουκρανία, τις πολιτιστικές και τις συσκευτικές διαφορές και τις εντάσεις που δημιούργησαν. Η προστασία των μειονοτήτων είναι βασικό θέμα. Θα πρέπει να προτάξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και θα πρέπει να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ο Γζιμπ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν ειδικό ρόλο για διαδραματίσει με ειδικέ ε, αρμοδιότητε και καθήκοντα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα ε, στη μη διάκριση, την ισότιμη μεταχείριση όλων, ε, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών και των παιδιών και των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στη βία. Ένα από τα πιο δικαι... σημαντικά δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην θρησκευτική ελευθερία και στην πολιτική διαφορετικότητα. Τα έχουμε αναφέρει όλα αυτά στα έγγραφά μα και στι αιτήσει εκθέσει για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και στι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαρκούν όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Γιατί πολύ συχνά στι χώρε ε, με τι οποίε έχουμε τέτοιε σχέσει, που είναι μάλιστα προνομιούχε, για παράδειγμα, χώρε με τι οποίε έχουμε υπογράψει συμφωνίε εταιρική σχέση, σύνδεση που έχουν λάβει αναπτυξιακή βοήθεια ή συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα συνεργασία. Σύμφωνα με οι πληροφορίε που λαμβάνουμε από ε, πολλού ε, οργανισμού ε, παρακολούθηση, όπως για παράδειγμα το Open Doors, η Βόρεια Κορέα παραμένει η χώρα που διώκει σε μεγαλύτερο βαθμό τους χριστιανούς. 100.000 χριστιανοί κρύβονται αυτή τη στιγμή και θεωρούνται εχθροί του κράτους. Ε, υπάρχουν πολλές ε, διώξεις και στις ε, χώρες της Σαχάρης Αφρικής, ιδίως στη Σομαλία. Παρότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις, παρόλα αυτά η Εκκλησία και πάλι κρύβεται και στο Πακιστάν έχουμε πολλά αρνητικά παραδείγματα. Τον, το, τελεσμα, το περασμένο φθινόπωρο σχεδόν 90 χριστιανοί δολοφονήθηκαν σε μία επίθεση στη Πάσοβα. Η δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής είναι άλλη μια χώρα που θεωρείται επικίνδυνη. Έχουμε ήδη συζητήσει τα όσα συμβαίνουν εκεί. Η ε, Συμμαχία Σάλα ασκεί τεράστια βία στον χριστιανικό πληθυσμό. Οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους ε, σε φυγή, αλλά ας μιλήσουμε και για την αραμαϊκή μειονότητα που ομιλεί τα αραμαϊκά από ε, την εποχή του Χριστού και μάλιστα πλέον οδηγούνται ε, στην εξάλληψη. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 50-18 εκατομμύρια χριστιανών που διώκονται, αλλά και άλλες θρησκευτικέ μειονότητες. Και αυτός ο κατάλογος δυστυχώς συνεχώς ε, αυξάνεται. Πρόσφατα είδαμε και είχαμε ενδείξει ότι και οι ε, Τατάροι της Κρυμαίας έχουν μπει σε αυτόν τον κατάλογο. Συνήθως μιλάμε για ε, δολοφονίες εξαιτίας της διαφορετικότητας, εξαιτίας ε, του γεγονότος ότι ανήκουν στη διαφορετική θρησκευτική μειονότητα. Ενώ πλέον μιλάμε για ε, μια πολιτισμική κληρονομιά μια ολόκληρη γενιά. Ευχαριστούμε. Το, το λόγο έχει ο κύριο Χάουιτ για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πλέον έχουμε αφοσιωθεί σε μια τέτοια συζήτηση ε, για την συμφιλίωση του σεβασμού προς ε, την πολιτισμική διαφορετικότητα ε, χωρίς να διακινδυνεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό παραμένει μια πρόκληση και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω κάποιε από τι διαφωνίε που έχουν εκφραστεί στο παρελθόν μεταξύ αριστερά και δεξιά να ξεπεραστούν και επικροτώ την παράγραφο 16 με τι ιδέε που προασπίζει. Ερασπίζουμε και την έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα πολιτισμικά δικαιώματα και άλλα και τις πολιτικές ε, και αστικές ελευθερίες και ελπίζω και η αυριανή ψηφοφορία να καταδείξει αυτό. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό που οι ηγέτες ε, Μεγάλου Βασιλείου και Γερμανίας ε, επέκριναν την αρχή της πολυπολιτισμικότητας, μια αρχή που πρέπει να υπερασπιστούμε. Μα ανησυχεί επίσης ότι η ομάδα ECR με τους Βρετανούς συντηρητικού ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία στην παράγραφο 7. Αν δεν στηρίξουν αυτό θα σημάνει μεγάλη ντροπή ε, και για τη φήμη της χώρας μου. Να το πω και αυτό. Χαίρομαι που υπάρχει η παράγραφος 30 που ε, επιβεβαιώνει την δέσμευσή μας για τη συμπερίληψη της ρήτρας ανθρωπινών δικαιωμάτων στις ε, συμφωνίες μας. Όμως αυτά, αυτές οι ρήτρες θα πρέπει, θα πρέπει να τις επικαλούμαστε σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι αδύνατον. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για την καταδίκη ε, της ε, δίωξης θρησκευτικών μειονοτήτων. Ευχαριστώ ε, και όσους έκαναν τις ε, τελευταίες τους ε, παρεμβάσεις σε αυτό το κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων και ευχαριστώ την κυρία Γιαννάκου. Εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια ήμουν εκπρόσωπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη ομάδα μου. Ευχαριστώ λοιπόν και τι ενώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τι οποίε συνεργάστηκα. Ο δικός μας υπεύθυνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, εκπώνησε και μία πολιτική ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Εγώ προσπαθώ και παλεύω για έναν καλύτερο κόσμο και ε, η ηθική είναι κάτι το οποίο με καθοδηγεί. Διακόπτεται το μικρόφωνο του ομιλητή. Συνεχίζει μια πολύ σαφής διάκριση μεταξύ σωστού και λάθους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σβένσεν για ένα λεπτό. Έχω ασχοληθεί με την πολιτική για 15 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια ήμουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από όλο αυτό το χρόνο έχω την αίσθηση ε, ότι κάποια πράγματα ε, ότι είναι μια θλιβερή αυτή τη στιγμή και ευχάριστη ταυτόχρονα γιατί δίνω την τελευταία μου ομιλία. Χαίρομαι που ήμουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 5 χρόνια, που είμαι μεταξύ σας, και θα έχω πολλές αναμνήσεις από το Κοινοβούλιο. Ένα Κοινοβούλιο που υπερασπίσεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ε, ανθρώπινες ελευθερίες. Συχνά λέμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε απλώς για αυτά τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε και κάτι και να πετύχουμε. Συχνά μιλάμε για την οικονομική ανάπτυξη και μου αρέσουν αυτά τα επιχειρήματα, τα σέβομαι απόλυτα κύριε Πρόεδρε. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να είναι σημαντικό για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για μας τους ευρωβουλευτές, το πιο σημαντικό από όλα είναι η δημοκρατία. Το να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, το να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη φυλή τους, τη θρησκεία τους και οποιοδήποτε άλλο πεπιθήσεων έχουν. Τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Να μην αρχίσω να παριθμώ τελικά, γιατί οποτεδήποτε απαριθμούμε κάτι, πάντα κάτι ξεχνάμε. Αλλά κάθε ένας να έχει την αξία του, την αξιοπρέπειά του και τα δικαιώματά του δεν τα δίνει κάποια κυβέρνηση όλα αυτά. Αυτά είναι εγγενή. Ε, τα έχουμε λόγω της ανθρώπινης φύσης μας. Και όπως είπαν πολλοί, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διώξεις, ειδικά διώξεις χριστιανών. Ε, διώκονται λόγω της πίστης τους. Υπάρχουν ε, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας λένε ότι το 80% των διωκόμενων διώκονται λόγω της χριστιανικής τους πίστης. Από ό,τι φαίνεται, Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διώκονται είναι χριστιανοί. Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να το πούμε αυτό. Να το πούμε, να το πούμε απερίφραστα. Να μην φοβόμαστε για την ταυτότητά μα. Εδώ μιλάμε για την αρχή του κράτου δικαίου, για την ελευθεροτυπία, την ελεύθερη γνώμη μα. Δεν υπάρχει καμία, κανένα μονοπόλιο για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει απερίφραστα να σηκωθούμε και να πούμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Οι ρίζε μα είναι στο χριστιανισμό. Το κληρονομήσαμε αυτό. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Και δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε να το λέμε. Γιατί μια και μιλάμε για την ανοχή, για την αποδοχή. Θα πρέπει να πούμε ποιε είναι δικέ μα οι αξίε. Έχουμε τη δική μα ταυτότητα, τι δικέ μα αξίε. Θα πρέπει να τι στηρίξουμε και να σεβαστούμε παράκλα τι ιδέε και την ταυτότητα των άλλων. Πρόεδρε, θέλω να σα πω ότι μια και είναι η τελευταία μου μιλή αυτή, η πιο ε, ακριβή μου επιθυμία είναι η ανθρώπινη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αυτή που θα καθοδηγεί το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ο κύριος Ζάλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς δεν Έχουμε καθήκον να υποστηρίξουμε μεμονωμένες θρησκείες. Έχουμε όμως το καθήκον να υποστηρίξουμε της, ε, την ύπαρξη των θρησκειών και το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Ο κοσμικισμός δεν σημαίνει πρέπει να είμαστε άθεοι, σημαίνει ότι πρέπει το κράτος να εξασφαλίσει την ελευθερία για όλες τις θρησκείες και όλες τις κοσμοθεωρίες. Είναι λοιπόν το καθήκον του κράτους να εξασφαλίσει αυτό το γεγονός και η κοινωνία των πολιτών επίσης θα πρέπει να το εξασφαλίσει. Για να είναι λοιπόν ελεύθερη θρησκευτική συνείδηση, το ίδιο το κράτος πρέπει να είναι κοσμικό. Πρέπει λοιπόν το κράτος να εξασφαλίσει αυτή την ελευθερία και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στην εξωτερική μας πολιτική. Η υπεράσπιση της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης και της δυνατότητας ακόμα να αλλάξει καλής θρησκεία αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε έξω ούτε μέσα στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι πολλοί θέλουν να επιβάλλουν ορισμένε αρχές όπως γίνεται στο Ουγγρικό Σύνταγμα. Αυτό είναι λάθος για μας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο σοβαρά φαινόμενα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, λέει ο κύριο Πόσελ. Το ένα φαινόμενο είναι η κατάχρηση της θρησκείας και η εκμετάλλευσή της. Το άλλο φαινόμενο είναι η καταδίωξη των θρησκειών και των ιερέων και η κατάλυση της θρησκευτική ελευθερίας. Όταν υπάρχει εκμετάλλευση της θρησκείας για ιδεολογικούς στόχους για να δικαιολογήσει βίαιους ή τρομοκρατικούς σκοπούς και όταν σκοτώνονται άνθρωποι καταδιώκονται στο όνομα της θρησκείας. Δεν υπάρχει μόνο ο Ισλαμισμός δυστυχώς. Έχουμε και άλλα φαινόμενα. Βλέπουμε αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Πούτιν ο οποίος απειλεί την Ευρώπη γιατί τώρα θεωρεί τον εαυτό του ως υπέρμαχο και προστάτη του χριστιανισμού. Αλλά είναι ένας μαζικός δολοφόνος και ένας επιθετικός ηγέτης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί προστάτης του χριστιανισμού. Έχουμε άλλα φαινόμενα, όπως η καταδίωξη ε, της θρησκευτική ελευθερίας και ιδίως των χριστιανών. Εδώ πρέπει η εξωτερική μας πολιτική να δράσει αποφασιστικά για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει σεβασμός στη θρησκευτική ελευθερία ανεξάρτητα από ποια θρησκεία πρόκειται. Στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρονται οι θρησκευτικές ρίζες της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πολυμορφία. Αλλά βλέπετε το καθεδρικό του Στρασβούργου σε αυτή την πόλη και βλέπετε ότι η Ευρώπη έχει σημαδευτεί από τον χριστιανισμό και από τον Ιουδαϊσμό. Αυτές είναι οι ρίζες της Ευρώπης και το κοσμικό κράτος δεν είναι ένα κράτος το οποίο κόβει αυτές τις ρίζες και τις αγνοείς. Ένα κοσμικό κράτος είναι ένα κράτος που δεν υποχρεώνει κανένα σε συγκεκριμένες θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Εμείς όμως κατά 80% είμαστε χριστιανοί στην Ευρώπη έχουμε αυτές τις βαθιές χριστιανικές ρίζες και γι' αυτό έχουμε μια ιδιαίτερη υποχρέωση να δράσουμε για να αποφύγουμε την καταδίωξη σχετικούς λόγους, ιδίως των χριστιανών, χωρίς να παραγνωρίσουμε και την αντίστοιχη καταδίωξη άλλων. Θα πρέπει προφανώς να εξασφαλίσουμε τον στόχο να υπάρχει θρησκευτική ελευθερία για όλους και ως χριστιανοί είναι πραγματικά καθήκον μας να το κάνουμε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η θρησκευτική ελευθερία. Αυτοί οι οποίοι θέλουν τη θρησκευτική ελευθερία δεν την περιορίσουν μόνο στον εαυτό τους. Μία θρησκεία υπερασπίζει όλες τις θρησκείες. Όποιος δεν σέβεται μία θρησκεία δεν σέβεται καμία. Αυτός ο οποίος σκέφτεται μόναχα τους δικούς του τη δική του θρησκευτική κοινότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να εξασφαλίσει <clears throat> την ειρήνη γιατί δεν θα έχει καταλάβει το ρόλο και τη σημασία των θρησκειών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να αγωνιζόμαστε για τη θρησκευτική ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μέρσκι δεν είναι παρόν και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, παρότι δεν υπάρχουν πολλοί παρόντες, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Η ελευθερία, η θρησκευτική και η αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά σήμερα. Καθώς προοδεύουμε και καθώς ε, η ανθρώπινη ράτσα έχει όλο και μεγαλύτερα επιτεύγματα. Κάθε πέμπτη το απόγευμα ε, συζητάμε αυτά τα θέματα, ε, εντοπίζουμε τις αδικίες σε όλο τον πλανήτη. Θα το ξανασυζητήσουμε και αύριο το απόγευμα λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα, ειδικά τις αδικίες που γίνονται στους χριστιανούς στο Πακιστάν πιο συγκεκριμένα. Και είναι σίγουρο ότι γίνονται τεράστιες αδικίες αντί των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Και εμείς, ειδικά στην ομάδα μας, όπως είπε ο κύριος Πόσελτ και άλλοι ομιλητέ, εμείς θα πρέπει να τους υπερασπιστούμε κυρίως. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε έτσι την ελευθερία όλων των θρησκειών και ακόμα και των άθεων που δεν πιστεύουν σε κανένα Θεό. Και αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα επόμενα πέντε χρόνια της επόμενης, δηλαδή, του επόμενου κοινοβουλίου θα ήθελα να δω το εξή να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές που έχουμε για την ανάπτυξη και την υποστήριξη χωρών και συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η θρησκευτική ελευθερία θα γίνει πραγματικότητα και σε αυτές τις τρίτες χώρες θα αναγνωριστεί η πολιτιστική ποικιλομορφία, τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί είναι σκανδαλώδες να βλέπουμε πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά ε, σε όλο πλανήτη ε, όπου οι γυναίκες είναι πολίτες δεύτερης κατηγορία ή δεν έχουν ε, κανένα δικαίωμα ή άνθρωποι που καταδικάζονται με την εσχάτη των ποινών, όπως είπαν διάφοροι συνάδελφοι. Δεν έχω κανέναν που ζητάει το λόγο στη διαδικασία του Catch the Eye, άρα ο κ. Κούρκουλα θα κάνει ελληνικέ παρατηρήσει. Ευχαριστώ επίσης ε, τους εξέτοιμου βουλευτέ για αυτή την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Θα μελετήσουμε βεβαίω με προσοχή το περιεχόμενο του ψηφίσματος ήθελα να παρατηρήσω ότι σε σχέση με τις ε, θρησκευτικές ελευθερίες βεβαίως η προστασία της ε, ελευθερίας της θρησκείας και η αποφυγή οποιασδήποτε βίας κατά των θρησκευτικών κοινοτήτων ε, είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες και στις κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες αναφέρθηκαν στην πρωτολογία μου. επίσης θέλω να ότι η η κυρία άστον και το συμβούλιο έχουν επανειλημμένα ε, άμεσα αντιδράσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καταπάτησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων ή άσκησης βίας ε, κατά θρησκευτικών κοινοτήτων αναφέρω ενδεικτικά το ιράκ το ιράν ε, δηλώσεις για την αλεξάνδρεια για το πακιστάν για την τινησία και βεβαίως για το δράμα το οποίο εκτελήσεται στη συρία και το οποίο πράγματι ε, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση ε, ιστορικές θρησκευτικές κοινότητες στη χώρα αυτή που υπήρχαν επί αιώνες. Είπα λοιπόν, όπως είπα, θα μελετήσουμε με προσοχή το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Ε, συμφωνώ απόλυτα και με αυτό που είπε η κυρία Γιαννάκου ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να επιβάλλει τους δικούς της πολιτιστικούς κώδικες σεβόμαστε την πολιτισμική πολυμορφία εξάλλου ο σεβασμός της πολιτισμικής πολυμορφίας αποτελεί και θεμελιώδη λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και στο εσωτερικό της ευρώπης. επιτρέψτε μου πριν κλείσω αυτή την παρέμβασή μου ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, βουλευτές που ασχολήθηκαν με το θέμα και κυρίως αυτούς για τους οποίους ε, αυτή η θητεία είναι η τελευταία. ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία γιαννάκου για την εξαιρετική πολυετή προσφορά της στην ευρωπαϊκή ενοποίηση η οποία είναι γνωστή ευρύτερα δεν θα τολμήσω να την απαριθμίσω τώρα γιατί θα χρειαζόμουν πολύ χρόνο απλώς να αναφέρω ε, πρόσφατα τον ε, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση ενός άλλου σημαντικού νομοθετήματος ε, στην υιοθέτηση του κανονισμού για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε γιαννάκου για όλη την προσφορά σας. τα τελευταία πολλά χρόνια έχετε νομίζω τέσσερις φορές εκλεγεί ευρωβουλευτής και σας εύχομαι καλή τύχη στις επόμενες δραστηριότητές σας. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Έχουμε ακόμα ε, μία πρόταση για τη συζήτηση. Λοιπόν, κλείνει εδώ πέρα η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Κυρίε και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημέρα διάταξη είναι η έκθεση SWAB. για τις ε, παραβάσεις του ε, δικαίου ανταγωνισμού. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Schwab.